God morgon allihopa. Jag eh, pratar svenska, så att om ni inte förstår det så föreslår jag att ni tar upp era hörlurar. I will speak Swedish. So. Λοιπόν, καλημέρα σας. Και θα σας δώσω, μια που μιλάω σου ειδικά, λίγα λευτερόλεπτα να βάλετε τα ακουστικά σας για να μπορέσετε να ακούσετε τη διερμηνία. Καλώ ήρθατε στη συνεδρίαση της Επιτροπής. Ξεκινάμε με το σημείο 1, υιοθέτηση της ημερήσια διάταξη. Δεν έγιναν προτάσεις για αλλαγέ και θεωρώ ότι εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη. Περνάμε στι ανακοινώσει του Προέδρου. Θα ήθελα να συγχαρώ τον συνάδελφο που ανέλαβε ένα αξίωμα στην Επιτροπή Άμυνας, τι τη συνάδελφο μάλλον, την Αρμέλ, είναι και εκείνη ευχαριστημένη, το ξέρω. Δεν χαίρομαι, Αρμέλ, που φεύγεις, αλλά χαίρομαι που αναλαμβάνεις αυτό το σημαντικό αξίωμα. Ξέρω πολύ καλά ότι και η Επιτροπή στην οποία πηγαίνει θα χαρεί να σε έχει. Εγώ ξέρω πολύ καλά ότι είσαι μια θαυμάσια συνεργάτη, πάντα δούλευε εξαιρετικά, μπορώ να το πω αυτό. Και πραγματικά πάντα ήσουν πολύτιμη και μας βοηθούσες σε όλα τα προβλήματα. Από μία μεριά λοιπόν θλίβομαι που φεύγεις, που αλλάζει υπηρεσία. Από την άλλη χαίρομαι που σου προέκυψε αυτή η ευκαιρία. Και χαίρομαι βέβαια που θα παραμείνει στο Κοινοβούλιο. Ωραία. Θέλω να καλωσορίσω έναν άλλο διοικητικό υπάλληλο που έρχεται στη δική μας επιτροπή, στο Policy Department. Καλώς ήρθατε και καλή δουλειά. Περνάμε τώρα στις ανακοινώσεις του Προέδρου σχετικά με τα πρακτικά και αν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις θεωρώ ότι εγκρίνονται. Θα πρέπει να εγκρίνουμε τα πρακτικά της 20 Απριλίου, 8 Μαρτίου, 10 Ιουλίου και ενδεκάτης, λέει ο Πρόεδρος, Οκτωβρίου. Προτείνω την υιοθέτησή τους. Πάμε στο σημείο 8. Προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων για την περίοδο 13-15 και παρουσίαση της έκθεσης ε, ανασκόπησης εφαρμογής του προγράμματος δράσης του Πεκίνου ε, από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελπίζω να γίνει μια ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων εδώ. Σε δύο εβδομάδες περίπου η Επιτροπή θα πάει στο Βίλνιους όπου θα συναντήσει τη μελλοντική Προεδρία του Συμβουλίου στο μέλλον θα υπάρχουν τακτικές επαφές. Θα το συζητήσουμε και στις συνεδρίες των συντονιστών. Και χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις, θέλω να δώσω το λόγο στον κύριο Λάμπακ, στην κυρία Λάμπακ. Ευχαριστώ και καλημέρα στα μέλη της Επιτροπής Γυναικών. Χαίρομαι που μας δίνετε την ευκαιρία να συζητήσουμε τις προτεραιότητές μας για τα επόμενα τρία χρόνια. Έχω μία παρουσίαση με διαφάνειες. Να σας πω καταρχάς τι κάναμε τα πρώτα δυόμιση-τρία χρόνια. Και θα σας παρουσιάσω επίσης και τι σκοπεύουμε να κάνουμε στο μέλλον, στο δεύτερο μισό του προγράμματος εργασίας. Σε δύο μέρες το Διοικητικό μας Συμβούλιο θα συναντηθεί και ελπίζουμε να υιοθετήσει το πρόγραμμα εργασίας του δεύτερου μισού της θητείας μας και συνεχεία θα τυπωθεί. Θα σας μοιράσουμε το πρόγραμμα. Να ξεκινήσουμε τα διοικητικά γιατί εκεί ήταν η μεγαλύτερη εστίαση τα πρώτα δυόμιση χρόνια. Γιατί το να ξεκινήσει μια υπηρεσία από το μηδέν πρέπει να προγραμματίσει τις πληρωμές, ε, τις διοικητικές δομές, τις οικονομικές δομές και αυτό χρειάζεται χρόνο. Πρέπει να το κάνουμε αυτό με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δεν είχαμε παρατηρήσεις για παρατυπίες ε, στους ε, οικονομικούς λογαριασμού. Αν δείτε τι έγινε το 2011 και το 2012, τη σύγκριση των δύο ετών, θα δείτε ότι βελτιώσαμε τις πληρωμές, δηλαδή αυτό που προγραμματιζόταν στο πρόγραμμα ε, δράσους, ε, από το 44 πήγε στο 64%, 65% και αυξάνεται. Ο στόχος είναι να φτάσουμε το 100%. Αν κοιτάξετε την εκτέλεση του προϋπολογισμού, τα πρώτα δυόμιση χρόνια, το 2010, όταν υιοθετήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο το πρόγραμμα εργασίας και αρχίσαμε να χρησιμοποιούμε τον, τον προπολογισμό για τον τίτλο 3 για την ισότητα των φύλων. Δεν είχαμε χρησιμοποιήσει όλο τον προϋπολογισμό ε, τώρα έχουμε πολύ μεγαλύτερη εκτέλεση μέσα στο 2012, όπου έχουμε ένα μικρό πλεόνασμα που θα μεταφερθεί την επόμενη χρονιά και αυτό είναι τρεις φορές μικρότερο σε σχέση με την πρώτη χρονιά. Τι καταφέραμε. Θέλουμε να βελτιωθούμε. Τον πρώτο φόνο ήταν αδύνατο να φτάσουμε στο establishment plan που ήταν στο δημοσιονομικό δελτίο. Τώρα έχουμε διάφορες εθνικότητες, δεν έχουμε και τις 27, έχουμε 19, είναι το 70% από όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για φυσικούς λόγους, οι περισσότεροι οργανισμοί που φιλοξενούνται στα κράτη-μέλη ε, δείχνουν αυτό το μοντέλο. Το διοικητικό τους προσωπικό είναι καταρχάς ε, ε, Λιθουανοί 21%. Μειώθηκε κατά 3% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Η συνεχεία είναι οι χώρες της Κεντρικής και Νότιας Ευρώπης, οι επόμενοι πολυεθνικότητες. Αν δείτε την ε, ισότητα, την ισορροπία των φύλων, προσπαθούμε να υπάρχει ισορροπία μεταξύ ανδρών και γυναικών. Αλλά δεν είναι εύκολο αυτό, γιατί δεν έχουμε πολλούς άντρες που ασχολούνται στην αγορά με τέτοια θέματα ισότητας των φύλων. Είναι το 1 τρίτο αυτή τη στιγμή οι άντρες. Το 2011 είχαμε μια μικρή αλλαγή μόνο. Η εξέλιξη του προσωπικού όπως βλέπετε, σε σχέση με το 2009, ή μάλλον το 2009, είχαμε λίγα μέλη στο προσωπικό. Ήμασταν στην αρχή. Βλέπετε πώς α, α, μεγάλωσε το προσωπικό, εξωτερικές και εσωτερικές κατηγορίες. Πέρα από, τους, από αυτούς που είναι σε μπλε, που είναι οι μόνιμοι, και έχουμε φτάσει στο 100%. Έχουμε και συμβασιούχου υπαλλήλου ανάλογα με τις διαθεσιμότητες του προπολογισμού και μπορούμε να τους προσλάβουμε για συγκεκριμένα ε, καθήκοντα. Έχουμε και αποσπασμένους ε, εθνικούς εμπειρογνώμονες. Είναι πολύτιμοι γιατί όχι μόνο ε, εκπροσωπούν τις παραδόσεις, την κουλτούρα και τις γνώσεις του συγκεκριμένου κράτους μέλους τους, αλλά επίσης τους προσλαμβάνουμε για συγκεκριμένα καθήκοντα και προς το παρόν οι περισσότεροι από τους αποσπασμένους εθνικούς εμπειρογνώμονες ε, ξέρουν θέματα που, γνωρίζουν θέματα που αφορούν τη βία ε, λόγω φύλου. Ασχολούμαστε με αυτά τα θέματα. Επίσης ε, έχουμε και μαθητευόμενους. Χαιρόμαστε για αυτή τη δυνατότητα γιατί είναι νέοι, γιατί έχουν καινοτόμα ματιά και έρχονται στο Ινστιτούτο μας, στον οργανισμό μας, ε, με τις γνώσεις τους, με την απόψή τους. Έτσι λοιπόν εξελίσσεται το προσωπικό μας. Όπως είπε και ο Πρόεδρος, με μεγάλη χαρά θα έρθει η αντιπροσωπεία το, της Επιτροπής Γυναικών ε, στα νέα μας γραφεία, μόνιμα γραφεία πια, που και είμαστε ο μόνος οργανισμός μέχρι στιγμή που έχει αυτό το μοναδικό συνδυασμό εκπροσωπήσεις ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μάλλον, έχουμε τα, τα ίδια γραφεία. Τα μοιραζόμαστε. Έτσι δηλαδή είμαστε και πιο αποτελεσματικοί με μικρότερο κόστος ε, και συνεργαζόμαστε και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Από την 7η Ιανουαρίου συμβαίνουν αυτά. Ε, από το τέλος του 2011, τι συνέβη. Υπογράψαμε μία συμφωνία με την κυβέρνηση της Λιθουανίας ε, για την έδρα υποχρεωτικό κομμάτι για την εγκατάσταση του οργανισμού και η συμφωνία αυτή προβλέπει κάποια επιπλέον δικαιώματα για το προσωπικό, για να προσελκύσουμε προσωπικό και να και άνθρωποι αυτοί να εγκατασταθούν στο Βίλνιους και για να ε, ενταχθούν πιο μαλά στην κοινωνία της Λιθουανίας. Η κυβέρνηση υποσχέθηκε να υποστηρίξει την δημιουργία του Ευρωπαϊκού Σχολείου, κάτι που συζητήσαμε με την κυβέρνηση. Το, τώρα, για την λειτουργία. Από το 2010 έχουμε συνεχή αύξηση του προσωπικού. Ξεκινήσαμε καταρχάς με το πρώτο μας καθήκον, την, πιο, την πρώτη μας αρμοδιότητα που είναι και, ήταν και πιο περίπλοκη. Υποστήριξη των Προεδριών του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αναθεώρηση της πλατφόρμας για δράσεις και είχαμε τέσσερις εκθέσεις και τέσσερα απορίσματα. Ε, ένα από αυτά τα έχουμε μοιράσει στους φακέλους σας, τα έχετε μπροστά στα καθίσματά σας. Οι τέσσερις εκθέσεις για την Πολωνική, Δανέζικη, Κυπριακή και Ιρλανδική Προεδρία δόθηκαν στις Προεδρίες του Συμβουλίου ε, με βάση τα συμπεράσματα με βάση τις οποίες ετοιμάστηκαν και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου. Λοιπόν, επίσης, για την Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάσαμε και τέσσερις νέους δείκτες για την... Ε, Εδώ δεν είχαμε στατιστικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να αναθεωρήσουμε τους ε, δείκτες για την κλιματική αλλαγή και τις ε, γυναίκες. Δηλαδή οι γυναίκες ε, στους τομείς λήψης των αποφάσεων και η αναλογία ανδρών και γυναικών στην εκπαίδευση σε επιστημονικούς και τεχνικούς τομείς. Τώρα έχουμε όλα αυτά τα στοιχεία στη βάση δεδομένων μας, υπάρχουν και προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την γνώση για τους δείχτες και να τη μοιράσουμε τα θεσμικά όργανα και στους οργανισμούς ε, που τα χρειάζονται, γιατί είναι σημαντικά, συγκρίσιμα και μπορούν ε, οι ενδιαφέρομενοι να βλέπουν τις αλλαγές. Επίσης, έχουμε νέες δέσμες σε συγκρίσιμο και αξιόπιστων δεδομένων για την κλιματική αλλαγή και για τον αριθμό και έκταση και χρήση των υπηρεσιών ε, που υπάρχουν στη διάθεση των γυναικών θυμάτων βίας. Αυτά τα βλέπετε στην έκθεση που σας μοιράσαμε σήμερα και στο, στην ιστοσελίδα μας. Τι βλέπουμε από τα διάφορα σχόλια στην ιστοσελίδα και στα κοινωνικά μέσα. Πολλοί οργανισμοί, πολλά άτομα και πολλά θεσμικά όργανα χρησιμοποιούν αυτή τη βάση δεδομένων για τις γυναίκες και άντρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση νούμερα και στοιχεία και συνεχώς αναθεωρούμε και επικαιροποιούμε τα δεδομένα, τόσο ώστε οποτεδήποτε υπάρχει ενδιαφέρον από οποιονδήποτε να χρησιμοποιεί αυτά τα, τα στοιχεία ε, για να ξέρει ποια είναι η κατάσταση και πώς απεικονίζεται σήμερα. Επίσης, ε, για την ίση εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών και την ισότητα των φύλων σε όλες τις, τις συμπερίληψη μάλλον αυτού του στοιχείου σε όλες τις πολιτικές. Ε, επιλέξαμε ένα εργαλείο από όλα τα διαθέσιμα και που ήταν η κατάρτιση των δύο φύλων. Είδαμε τι συμβαίνει σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Δημιουργήσαμε μια βάση δεδομένων για τους πόρους, για την κατάρτιση των φύλων. Έχουμε πάνω από 200, 200 πηγές από διάφορες γλώσσες. Ορισμένα στοιχεία αυτά, από αυτά χρησιμοποιούνται. Και όταν θέλουν τα θεσμικά όργανα να εξοικονομήσουν χρόνο και χρήμα, μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν. Ευχαριστούμε το Κοινοβούλιο που συμμετείχε στη διάσκεψη πέρυσι όταν συζητήσαμε τα θεσμικά όργανα, τα κράτη-μέλη, οι φορείς που παρέχουν κατάρτιση, οι ερευνητές, για το ποια είναι η αποτελεσματική κατάρτιση των δύο φύλων και ποια είναι τα κριτήρια για να χρησιμοποιήσουμε την κατάρτιση, ούτως ώστε να αφυπνίσουμε τον κόσμο για τη σημασία της ισότητας των φύλων, αλλά και για τη σημασία της σωστής κατάρτισης να το κάνουν. Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα είναι αυτό που θα, που θα συμβεί τον Ιούνιο. Είναι ο δείκτης για την ισότητα των δύο φύλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βασίζουμε τη δουλειά μας, τη δουλειά που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πρώτο δικό χάρτη όπου τα βασικά στοιχεία του δίκτυ είχαν ήδη συζητηθεί και υποστηρίζουμε τη στρατηγική της Κομισιόν για την ισότητα των δύο φύλων. Η Κομισιόν μας έδωσε αυτό το καθήκον να το κάνουμε και τώρα ετοιμάσαμε ένα μοναδικό προϊόν. Είναι η πρώτη φορά δηλαδή που αυτός ο δείκτης θα μιλάει για τις πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης και μόνο. Αναλύσαμε όχι μόνο την Ευρώπη 2020, αλλά και όλες, δηλαδή το γνωρίζονται αυτό, αλλά και όλες τις πολιτικές, για να δούμε ποιες από τις πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης κερδίζουν, θα κέρδιζαν από το να υπήρχαν ε, συγκεκριμένοι δείχτες που να αφορούσαν την ισότητα των δύο φύλων. Στις 13 ε, Ιουνίου, στις Βρυξέλλες, θα ξεκινήσει στις Βρυξέλλες με τη συμμετοχή της Επιτροπής ε, Γυναικών η παρουσίαση αυτού του προϊόντος, αυτού του δείκτη δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα σας στείλουμε και περισσότερες πληροφορίες αργότερα, αλλά βλέπετε όλους τους δείκτες που συνδέονται με διάφορες πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνόψισα λοιπόν αυτά τα οποία κάναμε αυτά τα δυόμιση χρόνια και έτσι ε, παρουσιάσαμε ε, ενημερωτικά φυλάδια γεμάτα με πληροφορίες και στοιχεία γύρω στις 160 σελίδες. Επίσης κάναμε έξι μελέτες για την βία κατά των γυναικών, βία που βασίζεται δηλαδή στη διάκριση του φύλου. Έχουμε νέα ε, στοιχεία, νέες τράπεζες δεδομένων και συνεργαζόμαστε με όλους τους συναφείς οργανισμούς για το, την ισότητα των φύλων, πολιτικές, οι καινούργιες μας τράπεζες δεδομένων έχουν, ας πούμε, συλλέγουν στοιχεία ε, υπό, τα κεφάλαια πολιτικές, ε, νομικά έγγραφα, μέθοδοι, ε, μέσα και καλές πρακτικές και ε, ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών. Αυτές, αυτά είναι τα στοιχεία που συλλέγουμε. Επίσης, ο αντιπρόεδρος, η αντιπρόεδρος Vivian Redding στην συζήτηση στρογγυλής τραπέζης στις 6 Μαρτίου παρουσίασε αυτή την ε, μελέτη την οποία κάναμε για την ε, γυναική, για την κλειτορίδο τομή και ε, Είμαστε έτοιμοι να υποστηρίξουμε την Κομισιόν σε περαιτέρω βήματα για αυτό το θέμα. Και αυτό αποτελεί λοιπόν μέρος του προγράμματος εργασίας. Επίσης έχουμε συζητήσει το θέμα του γυναικείου ακροτηριασμού της ε, κλειτοριδεκτομής και έχουμε οργανώσει και μία παρουσίαση η οποία θα συνοδευτεί από τα, την τεκμηρίωση που θα έχουμε έτοιμη. Όπως σας είπα υπάρχει και αυτή η τράπεζα δεδομένων στο διαδίκτυο, αλλά για κάθε κράτος μέλος προετοιμάσαμε ε, ένα φυλάδιο με τα στοιχεία, με τα δεδομένα τα οποία θα είναι διαθέσιμα για να μπορείτε να έχετε μια γενική άποψη, μια ανασκόπηση όλων των στοιχείων, τα, τα, τα, τα στοιχεία τα οποία έχουν καταγραφεί, τα νομικά έγγραφα και γενικά όλα τα δεδομένα και αυτά τα στοιχεία μπορούν να υποβληθούν ανα πάσα στιγμή διότι υπάρχουν στη γραμματεία της Επιτροπής μας και είναι στη διάθεσή σας όποτε θέλετε. Επίσης, πέρσι ένα άλλο περίπλοκο έργο που αναλάβαμε είναι το Κέντρο Τεκμηρίωσης και Αναζήτησης Πηγών. Εκεί συλλέγουμε όλη την, ε, τις γνώσεις, όλα τα μέσα, όλα τα εργαλεία τα οποία χρειαζόμαστε σε διάφορα επίπεδα. Ε, μας δόθηκε λοιπόν η εντολή να συγκεντρώσουμε όλες τις επιγές και όλη την τεκμηρίωση σε ένα κέντρο. Μέσω αυτού του κέντρου λοιπόν όλοι εσείς οι ερευνητές, οι ενδιαφερόμενοι, τα ε, οι διαφοράμενοι οργανισμοί, σύλλογοι και ενώσεις μπορούν να αποτανθούν σε αυτή την τράπεζα δεδομένων για να επιταχύνουν το έργο τους και να λαμβάνουν όλες τις προφορίες. Είναι στο διαδίκτυο. Έχουμε πάνω 170.000 εγγραφές διαθέσιμες στο διαδίκτυο. Δεν είναι αυτά τα οποία μαζεύουμε εμείς, αλλά συλλέγουμε. Είναι ένα συλλεκτικό κέντρο το οποίο εμείς διαθέτουμε και εκεί έχω συλλεγεί και εγγραφεί όλες οι πληροφορίες οι οποίες είναι χρήσιμες για τους ερευνητές. Επίσης έχουμε τώρα 26.000 εγγραφές ε, στο διαδίκτυο για την βία η οποία συνδέεται με τη διάσταση του φύλου και αυτά τα πέντε ευρωπαϊκά μεγάλα κέντρα τεκμηρίωσης χρησιμοποιούνται ως ε, κόμβι επαφής ε, για τη συλλογή και χρησιμοποίηση όλων αυτών των στοιχείων. Και κάτι άλλο το οποίο έχουμε επίσης ε, αποφασίσει και θα αρχίσει να υλοποιείται αυτό το έτος είναι το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Ισότητα των Φύλων, το Eurogender gender. Και πέρσι το παρουσιάσαμε σε μία από τις ε, συνεδριάσεις της Επιτροπής. Είχαμε ανακοινώσει λοιπόν τι θα γίνει αυτό και το, τα στελέχη μας το, το, το παρουσίασε. Αυτό το Eurogender λοιπόν θα χρησιμοποιηθεί για συζητήσεις για την ανταλλαγή πληροφοριών ακριβώς για αυτό το θέμα της ισότητας των φύλων και ε, θα γίνουν, θα οργανώσουμε πολλές συζητήσεις και στο διαδίκτυο αλλά και με επαφή με πολιτικούς θα καλέσουμε διάφορα προσωπικότητες για να μας εξέσουν τις απόψεις τους σε συγκεκριμένους τομείς. Και επίσης ε, εμπειρογνώμονες που θα μπορέσουν να μας παρουσιάσουν επιχειρήματα και να στηρίξουν την απόφαση αυτή που λάβαμε. Επίσης είμαι ευτυχής να σας πληροφορήσω ότι παρόλο που είναι μικρό και νέο το στοιχείο αυτό, ε, τα καταφέρουμε πάρα πολύ καλά με τα κοινωνικά μέσα επαφής. Είμαστε υπαρισμόν τέσσερα όσον αφορά τον αριθμό των ε, μελών μας στα διαδικτυακά κέντρα, κοινωνικά κέντρα και έχουμε συνδεθεί με όλους τους ε, φορείς που ασχολούνται με τα θεμελιώδη δικαιώματα κλπ. Είμαστε λοιπόν οι πρώτοι από, τις νέες, από τα νέα ιδρύματα, τις νέες υπηρεσίες, οι η οποία έχει τώρα την τέταρτη θέση όσον αφορά τον αριθμό φίλων και ατόμων που παρακολουθούν, μας παρακολουθούν. Επίσης, ε, τώρα ε, θέλουμε να παρακολουθήσουμε τον τρόπο εργασίας για το θέμα της ε, ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και θέλουμε να παρακολουθήσουμε τι ρόλους ε, τι ρόλους μοντέλα, ποιο είναι το προφίλ δηλαδή το οποίο πρέπει να παρακολουθήσουμε, να, να, σημειώσουμε ε, στο θέμα αυτό της διάσταση των, των φύλων. Ποια, ποια ακριβώς ε, είναι η ρόλη μοντέλα στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτά έχουμε κάνει συνοπτικά και θα ήθελα να σας ε, πω ότι το πρόγραμμα αυτό εργασίας, ε, το καινούριο, θα συνεχίσει την, ε, την πάνω στα θέματα αυτά, θα, θα διευρυνθούν βεβαίως οι τράπεζες δεδομένων, αλλά θα εστιάσουμε το καινούριο πρόγραμμα στην εδραίωση συνεργασίας διαφόρων δικτύων συνεργασίας και στην παγίωση του δίκτυου συνεργασίας με όλους τους συναφείς οργανισμούς και τα Ινστιτούτα που μπορούν να μας βοηθήσουν ε, και να τους βοηθήσουμε εμείς στη βελτίωση των εργασιών τους. Σας είπα λοιπόν ότι μετά από τρία χρόνια θα δούμε πώς ε, η εργασία την οποία κάνουμε εμείς έχει επηρεάσει την, ε, τη λήψη των αποφάσεων ε, στα θέματα αυτά γενικά. Θέλουμε λοιπόν να έχουμε, να, να μπορούμε να παρουσιάσουμε αξιόπιστα και σύγχρονα επίκαιρα στοιχεία για να δούμε πού υπάρχουν κενά, πού υπάρχουν προβλήματα θα εργαστούμε στην επικαιροποίηση της ε, ατζέντα για την ισότητα των φύλων. Κάθε χρόνο ανανεώνουμε αυτήν την ατζέντα για να μπορούμε ακριβώς να επισημάνουμε συγκεκριμένους τομείς οι οποίοι χρειάζονται μελέτη, οι οποίοι χρειάζονται δράση. Εκεί δηλαδή όπου υπάρχουν αδυναμίες, εκεί όπου δεν υφίσταται, εκεί που υπάρχουν μεγάλα προβλήματα στο θέμα της ισότητας. Και ενσωματώνουμε συνεχώς καινούργια στοιχεία. Έχουμε και ένα άλλο πρόγραμμα στο μεσοπρόθεσμο, ε, διευρύνουν ε, δηλαδή τι δραστηριότητε μας ε, και από απόψε συλλογή στοιχείων στο θέμα της βίας κατά των γυναικών και συνεργαζόμαστε και με το Κοινοβούλιο σε αυτό το θέμα και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε στο θέμα της διάστασης του φύλου και το να περιλαμβάνεται το θέμα αυτό σε κάθε πολιτική που εκπονείται. Είναι μια πολύ αποδυτική εργασία για μας. Και σε ένα νέο τομέα θα προσπαθήσουμε να αναπτύξουμε αναλυτικά μέσα, αναλυτικά εργαλεία, τα οποία θα μπορούν συνοπτικά να παρουσιάζουν τα ωφέλη ε, της ισότητας των φύλων ένα δίκτυ λοιπόν με μέτρησης των ε, πλεονεκτημάτων και των ωφελημάτων από τη διάσταση του φύλου. Θα συνεχίσουμε ε, να εδραιώνουμε την ε, καταγραφή και την αρχιοθέτηση στο Ινστιτούτο των Πολιτικών και των Μεθόδων Υλοποίησης που σημαίνει ότι οποιοδήποτε κράτο ή πολιτικό κόμμα θέλει να εξετάσει τι έχουμε κάνει στο παρελθόν κτλ. Όλα αυτά είναι καταγεγραμμένα. Και πρόσθετες δραστηριότητες, όπως σας είπα, έχουν δείξει τα πρώτα δυόμιση χρόνια, έχουν πάρα ε, μας έχουν εφολίσει πάρα πολύ σε όλα τα θέματα που μελετάμε. Συνεργαστήκαμε και με όλες τις χώρες οι οποίες ήταν ε, υποψήφιες προς ένταξη με τη Γενική Διεύθυνση Διεύρυνσης και διευρύναμε γενικά τους στόχους μας αυτά τα πρώτα τρία χρόνια. Αυτά έχουμε κάνει λοιπόν μέχρι σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Good morning, dear Καλημέρα σας, ε, αγαπητέ Πρόεδρε και μέλη της Επιτροπής. Ξέρω ότι μας πιέζει λίγο χρόνος για την παρουσίασή μου, αλλά ε, χαίρομαι ιδιαίτερα που έχετε ένα, μία έκθεση για την υποστήριξη των θυμάτων στο θέμα της ε, βίας κατά των γυναικών. Οπότε, εφόσον υπάρχει αυτή η έκθεση, θα τονίσω ή μάλλον θα συνοψίσω τις πληροφορίες που θα βρείτε σε αυτήν την έκθεση για την υποστήριξη, στήριξη θυμάτων. Δεν θα επισέλθω σε περισσότερες λεπτομέρειες γιατί μπήκε στην ατζέντα, αλλά ήταν ένα από το θέμα το οποίο ήταν στην ατζέντα της Κυπριακής Προεδρίας και αποφάσισαν ότι στο ευρύ θέμα της βίας κατά των γυναικών θέλουν να προσέξουν περισσότερο, την, ιδιαίτερα μάλλον, την στήριξη, την υποστήριξη που παρέχεται στα σήματα οι ορισμένοι δείκτες έχουν ήδη οθετηθεί από τη Δανική Προεδρία του 2002. Οπότε και το ε, πεδίο ισχύω των δικτών είναι πολύ ευρύ. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να παρουσιάσουμε μία ανασκόπηση της, ε, των αποτελεσμάτων όλων αυτών των δικτών που χρησιμοποιήσαμε. Και θα δείτε και στο έγγραφο που έχετε ότι το φάσμα των υπηρεσιών που αναθεωρήσαμε, που ερευνήσαμε και καταγράψαμε καλύπτει 13 κατηγορίες. 13 υποδείκτες. Είναι ευρείες αυτές οι 13 κατηγορίες. Αλλά η μεγαλύτερη χρησιμότητα της μελέτης είναι η εξής είναι η πρώτη φορά που συλλέξαμε στοιχεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο ε, για τις ε, υπηρεσίες αυτές. Ε, ξέραμε ότι οι κυβερνήσεις των κρατών μελών δαπανούν πολλά κονδύλια για αυτό το θέμα, αλλά δεν είχαμε συγκεκριμένες πληροφορίες ε, για τις συγκεκριμένες υπηρεσίε που χρηματοδοτούνται. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο στην καταπολέμηση της βίας των γυναικών εξετάσαμε το θέμα αυτό υπό τη σκοπιά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, και αυτό το στοιχείο θα το βρείτε και στα συμπεράσματα του Συμβουλίου. για να αποσαφηνίσω αυτά που κάνουμε. Εμείς επικεντρώνουμε την προσοχή μας στην βία στο σπίτι, στην, ε, στην οικιακή βία κατά των γυναικών εντός του σπιτιού. Ε, δεν είναι δυνατόν να ερευνήσουμε και να καταγράψουμε βία κατά των γυναικών σε όλους τους τομείς, ένα ευρύτερο το φάσμα. Κάνουμε μία διάκριση λοιπόν επίσης ε, μεταξύ των γενικών υπηρεσιών υποστήριξης θυμάτων και των ειδικών υπηρεσιών. Ε, εδώ θέλαμε ακριβώς να ε, καταγράψουμε τις διαφορές. Υπάρχουν οι υπηρεσίες που είναι γενικές για υποστήριξη θυμάτων, αλλά εμείς θέλαμε να δούμε ποια είναι τα προβλήματα τα συγκεκριμένα στην υποστήριξη γυναικών και παιδιών που είναι σήματα της βίας. Βεβαίως όλες αυτές οι πληροφορίες υπάρχουν, ε, ήθελα να παρουσιάσω και μερικές διαφάνειες. Θέλω να τονίσω ότι η έκθεση αυτή καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ε, και ε, στα κράτη-μέλη και ε, η μελέτη αυτή ασχολήθηκε και με την εγκληματικότητα και με τους δράστες και με τις αξιόπινες πράξεις. Ε, πραγματικά προσπαθήσαμε στο επίπεδο των κρατών μελών να συγκεντρώσουμε τα, όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία για το τι συμβαίνει Ε, επίσης κάναμε μία αξιολόγηση της ποιότητας των δεδομένων, ε, κάναμε μία ε, αξιολόγηση των ε, συντρόφων ή των ανθρώπων που ζουν με αυτές τις γυναίκες πάντων και αδικοπραγούν και με τα στοιχεία που συλλέξαμε Α, σε, καλύπτουμε και ακαδημαϊκές, ε, ακαδημαϊκούς, ε, ε και πανεπιστημιακά ιδρύματα. Επίσης ήθελα να προσέξω ότι υπάρχουν ορισμένες υπηρεσίες στην Ευρώπη που είναι ολο, ολοκληρωμένες και δεσπόζουσες όμως αλλού υπάρχουν μεγάλα ελλείμματα. Παραδείγματο χάρη υπάρχουν ειδικέ υπηρεσίες για την υποστήριξη γυναικών από ευάλωτες ομάδες, παραδείγματος χάρη μετανάστριες. Εδώ λείπουν στοιχεία, έχουμε πολύ λίγα στοιχεία από κράτη-μέλη, τι γίνεται με την παροχή υπηρεσιών υγείας, τι γίνεται με, την, με τις άδειες εργασίες κλπ. Κάνουμε τα πρώτα βήματα λοιπόν συλλογής των στοιχείων για τέτοιες ειδικέ ομάδες. Επίσης όσον αφορά ε, τα κράτη-μέλη πριν ή μετά, τι διεύρυνση. Τα περισσότερα στοιχεία τα έχουμε από τα παλαιότερα ε, κράτη-μέλη, πρώτης διεύρυνσης ε, δηλαδή, ε, όπου οι υπηρεσίες προστασίας ή ενασχόλησης με θέματα όπως η βία κατά των γυναικών ήταν πολύ πιο ανεπτυγμένες. Πρώτο 2004 λοιπόν. επίσης, έχουμε εδώ στην έκθεση πληροφορίες για το νομικό δίκτυο, για την νομοθεσία και πόσες χώρες καλύπτουν την υποστήριξη των γυναικών και τις παρεχόμενες υπηρεσίες, ε, counseling και παροχή ειδικών τηλεφωνικών γραμμών κτλ. Από, ε, ε, καλύπτουν δηλαδή όλες αυτές τις υπηρεσίες βάσει της νομοθεσίας. Πολλές φορές αυτές οι υπηρεσίες δεν είναι υποχρεωτικές, δεν ορίζονται από το νόμο και μπορεί να είναι πολύ προβληματική η, η, λειτουργία και η εδραίωσή τους. Το Συμβούλιο το Δεκέμβριο του 2010 υιοθέτησε συμπεράσματα επί τη βάση ε, της, των προτάσεων της Κυπριακής κυβέρνησης. Δηλαδή δέχτηκε τις προτάσεις μας και τις συστάσεις μας η Κυπριακή Προεδρία και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου αντανακλούν ακριβώς αυτές τις προτάσεις μας. Εμείς είπαμε ξεκάθαρα ότι η, η βία στο σπίτι είναι ε, ε, εμπίπτει σαφώς στον ποινικό κώδικα, στην ποινική νομοθεσία και και θα πρέπει όλες οι μορφές της βίας να καταδικαστούν ε, και να θεωρούνται ως ποινικά αδικήματα κατά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είπαμε λοιπόν ότι χρειάζονται, χρειάζεται περισσότερο συντονισμός ε, μεταξύ των εθνικών προγραμμάτων των κρατών μελών. Ε, επίσης, μόνο 15 κράτη έχουν νομικές διατάξεις ε, οι οποίες καλύπτουν τους δράστες της οικιακής βίας και τονίσαμε και την ανάγκη ε, ειδικών ε, υπηρεσιών, υπηρεσιών που θα έχουν συγκεκριμένου στόχους δηλαδή. Και αυτό θα αναφέρεται και στα συμπεράσματα του Συμβουλίου πόσο σημαντικό είναι να εφαρμόζεται η διάσταση του φύλου σε όλες αυτές τις προτάσεις. Υπάρχει και η νέα οδηγία που θα ορίζει τα ελάχιστα standards για τα δικαιώματα προστασίας των θυμάτων διότι δεν είναι σαφές το, το ε, γενικά το επίπεδο των δικαιωμάτων προστασίας αυτών των θυμάτων και, και ε, τι δικαιώματα έχουν. Όσον αφορά τη χρηματοδότηση, όλα αυτά υπάρχουν μέσα στην έκθεσή μου. Και ε, θα ήθελα να σταματήσω εδώ για να κάνω μία τελευταία παράκληση, να διαβάσετε ενδελεχώς την έκθεση αυτή που παρέχει όλες αυτές τις πληροφορίες. Ευχαριστώ τις δύο μελίτες. <clears throat> Και επειδή και ευχαριστώ επίσης, λέει ο Πρόεδρος, που μας δώσανε μια εμπρεστατωμένη εικόνα των δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου αυτού, ξεκινώντας από την πλατφόρμα του Πεκίνου. Είναι σημαντικό να δούμε. Να δώσω πρώτα το λόγο στην κυρία Μπάουερ. Uh, ευχαριστώ πολύ. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η παρέμβασή σας. Μας μιλήσατε για αυτή την πολύ μεγάλη δουλειά που έχει κάνει το Ινστιτούτο σας. Και το πιο σημαντικό που κάνατε είναι ότι καταφέρατε να βρείτε μια θέση στον ήλιο και μια στέγη πάνω από τα κεφάλια σας. Και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Χαίρομαι γιατί έκλεισε αυτό το πρώτο κεφάλαιο της ιστορικής σας διαδρομής. Και τώρα βλέπουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Όμως, την περασμένη εβδομάδα κάναμε μια συζήτηση για διάφορα θέματα που αφορούν τις γυναίκες στην Ολομέλεια και κάποιος, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς ποιος, ρώτησε το εξής. Τι κάνει το ΕΙΚΕ, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων, μα είναι αόρατη. Τέθηκε λοιπόν αυτή η ερώτηση. Η γραμματεία σας ίσως θα πρέπει να το εξετάσει αυτό. Τι μπορείτε να κάνετε για να αυξήσετε την ορατότητά σας. Να μην αντιμετωπίσετε συνεχώς αυτή την απειλή συγχώνευσης μεταξύ των Ινστιτούτων. Δεν ήταν δύσκολη διαδικασία έγκρισης ε, της ε, δημιουργίας αυτού του Ινστιτούτου. Ορισμένοι το θυμόμαστε καλά αυτό, δεν ήταν καθόλου εύκολο. Θα ήθελα το ΕΙΚΕ, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων, να εμπλακεί περισσότερο στη δική μας δουλειά. Για παράδειγμα, του χρόνου στις 8 Μαρτίου θα μπορούσαμε να έχουμε κάποιο δίκτυ για την ισότητα των φύλων. Υπάρχουν πολλά που μπορούμε να κάνουμε. Πολλά μπορείτε εσείς να κάνετε για να μας βοηθήσετε οι δικές σας γνώσεις μας είναι εξαιρετικά χρήσιμες. Για παράδειγμα, αυτό που κάνετε για τις προεδρίες. Συνήθως, εμείς σχεδιάζουμε τις επισκέψεις μας στην εκάστοτε Προεδρία. Εάν ξέρουμε εκ των προτέρων ότι έχετε κάνει δουλειά για αυτούς, αυτό είναι χρήσιμο πολύ για όλους μας. Νομίζω λοιπόν ότι πάρα πολλές διαστάσεις δεν έχουν εξερευνηθεί ακόμα. Υπάρχουν πάρα πολλά σημεία που μπορούμε να αναπτύξουμε έτσι περαιτέρω για να βελτιώσουμε τη συνεργασία μας. Και θα ήθελα και να θέσω και ένα άλλο ερώτημα που έχει να κάνει με την άλλη πλευρά του νομίσματος. Ο δείκτης ε, για την ισότητα των φύλων περιλαμβάνει και την πρόσβαση σε νομικά μέσα επανόρθωσης. Είναι ιδιαίτερο κάπως το ζήτημα αυτό και συχνά το λησμονούμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, καλό θα ήταν να ακούσουμε δύο ερωτήσεις πριν δοθούν οι απαντήσεις. Πρώτα η κυρία Πέρες και μετά η κυρία Κλιβέτη. Ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομη. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τις παρουσιάσεις σας για τη δουλειά του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων. Αναμφισβήτητα θα μας χρησιμεύσουν ιδιαίτερως στη δική μας δουλειά εδώ στην Επιτροπή για τις Γυναίκες και την Ισότητα των Φύλων. Ως εκπρόσωπος της ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών θέλω να πω ότι μας ικανοποιεί ε, το γεγονός ότι το Ινστιτούτο πραγματικά φέρνει αποτελέσματα, γιατί εμείς πιστεύαμε σε αυτό το Ινστιτούτο εξ αρχής και αποτελούσε αίτημα και διεκδίκησή μας να δημιουργηθεί ένα τέτοιο Ινστιτούτο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να έχουμε έγκυρα στοιχεία, πιστοποιημένα στοιχεία, για να μπορέσουμε να κάνουμε μια σωστή ανταλλαγή καλών πρακτικών. Σα συγχαίρω λοιπόν για τη δουλειά, της, για τη σας. Από εκεί και πέρα, το σημαντικό τώρα είναι ποιο ο καρπός της δουλειάς σας να χρησιμεύσει όχι μόνο για τις ενδιαφερόμενες, τις γυναίκες, για τους ανθρώπους, αλλά και για τους πολιτικούς ηθήνοντες, για τα θεσμικά όργανα, για τους φορείς, για να είναι χρήσιμα τα αποτελέσματα της δουλειάς σας για όλα τα κινήματα που εργάζονται υπέρ της ισότητας των φύλων και ε, υπέρ της καταπολέμησης της βίας εναντίον των γυναικών. Θα έπρεπε να έχουμε διάδοση όλων αυτών των αποτελεσμάτων στην οργανωμένη κοινωνία των πολιτών για να μπορέσουν οι γυναικείες οργανώσεις να βελτιώσουν τον τρόπο εργασίας τους ε, όταν δραστηριοποιούνται σε αυτό το τομέα. Ευχαριστώ πολύ. Τελευταία ερώτηση, κυρία Κλιβέτη. Πολύ σύντομα. Ε, θα ήθελα να μιλήσω γαλλικά γιατί είναι και η εβδομάδα της γαλοφωνίας. Ε, αυτή, αυτή η εβδομάδα. Να συγχαρώ λοιπόν την πρόεδρο του Ινστιτούτου και να πω ότι είναι γεγονός ότι η έκθεση της οποίας ε, ήμουν εισηγήτρια έδωσε λαβή για πάρα πολλά σχόλια για την απαλλαγή τελικά του ε, Ινστιτούτου. Το σημερινό ζήτημα είναι πολύ σημαντικό και έρχεται παράλληλα με το πρόσφατο μανιφέστο της ομάδας των σοσιαλιστών, το οποίο περιλαμβάνει αναφορά στην καταπολέμηση της βίας εναντίον των γυναικών. Πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε μαζί. Κάνετε πολύ καλή δουλειά και είστε πολύ χρήσιμοι ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Η Επιτροπή ενδεχομένως θα ήθελε να κάνει κάποιες παρατηρήσεις εν συντομία παρακαλώ. Ναι, πολύ σύντομα, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγχαίρει το Ινστιτούτο για τη δουλειά που έχει ε, επιτύχει τα τελευταία χρόνια. Πράγματι, βλέπουμε τώρα τα αποτελέσματα και αυτό είναι κάτι που το αντιληφθήκαμε όλοι μετά από αυτές τις δύο παρεμβάσεις. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ γιατί πράγματι ήσασταν σύντομος. Να δώσω τώρα το λόγο στις ε, δύο ομιλήτριες και σας ζητώ συγγνώμη γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο για τη συζήτηση. Σε κάθε περίπτωση ε, η παρατηρήσεις σας για τις ερωτήσεις που σας τέθηκαν μας ενδιαφέρουν ιδιαιτέρως. Ναι, θα είμαι σύντομη. Μιλήσαμε για την ορατότητα, είναι γεγονό αυτό. Έχουμε τώρα την πρώτη πρόταση για το πώς θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό θα είναι και το θέμα της συνεδρίασης των συντονιστών σήμερα. Και κάθε άλλη ιδέα είναι σημαντική για εμάς, γιατί εσείς ξέρετε τι πραγματικά χρειάζεται και όταν μας το λέτε εμείς βρίσκουμε τρόπους να το πετύχουμε. Τώρα, ως προς τις οργανώσεις ε, της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών, τις διάφορες κοινωνικές οργανώσεις και ούτω καθεξής. Πρώτη, πρώτο στρώμα επαφής είναι το ευρωπαϊκό επίπεδο. Το λόμπι του Ευρωπαϊκού των Γυναικών έχουν ένα φόρουμ πρόσβασης και έχουμε και μια μεγάλη συνάντηση στα τέλη Μαΐου και εκεί θα ε, τελειοποιήσουμε τη συνεργασία μας. Επίσης, η κοινωνική πλατφόρμα είναι μέλη του Φόρουμ των Εμπειρογνωμόνων. Θα συναντηθούμε και με αυτούς σήμερα. Και επίσης δουλεύουμε σε επίπεδο δικτύωσης. Θέλουμε να εμπλακούν διαφορετικές οργανώσεις. Φυσικά πρόβλημα είναι η γλώσσα. Δεν έχουμε προσωπικό που να μιλάει όλες τις γλώσσες. Και στις ε, οργανώσεις αυτές ενδεχομένως ε, μιλούν διαφορετικές γλώσσες και δεν μιλούν όλοι αγγλικά. Σε κάθε περίπτωση κάνουμε το πάνω για να προοδεύσουμε και να υπάρξει πρόεδρος, πρόοδος. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ διότι ήρθατε εδώ για να μας ενημερώσετε για τις δραστηριότητές σας. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσες οι παρουσιάσεις σας. Επίσης, θέλω να ξέρετε ότι θα συνεχίσουμε να συναντιόμαστε και θα διατηρήσουμε ανοιχτό αυτό τον διάβλο επικοινωνίας. Για άλλη μια φορά σας ευχαριστώ που ήρθατε στην Επιτροπή μας. Τώρα θα ξεκινήσουμε τις ψηφοφορίες. Πριν το κάνουμε, να ρωτήσω το εξής. Μπορείτε να μην κάνετε πάρα πολλά σχόλια κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, γιατί αυτό με δυσκολεύει ε, στη δουλειά μου. Δυσκολεύομαι να προεδρεύσω. Εάν θέλετε να κάνετε σχόλια, εάν θέλετε να επαληθεύσετε, αν υπάρχει κάτι που πιστεύετε ότι κάνω λάθος, τότε πραγματικά να το πείτε. Αλλά όχι άλλες απαρατηρήσεις αν έχετε την ευγενή καλοσύνη, γιατί ε, δυσχεραίνει πολύ το, το έργο μας. Αυτό ήθελα να σας πω. Ευχαριστώ λοιπόν γι' αυτό. Ξεκινάμε με το σημείο 9 τα δικαιώματα των γυναικών στις ε, χώρες υποπροσχώρηση των Βαλκανίων. Η συγγήτρια ενδεχομένω θα ήθελε το λόγο. Εν συντομία κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους και συγγητέ και και συγγήτριες για ε, τη συνεργασία τους. Πιστεύω ότι μετά από αυτή την ψηφοφορία θα έχουμε μια θαυμάσια έκθεση ε, πάνω στην οποία μπορούμε να στηριχθούμε κάθε φορά που θα έχουμε επαφή με τις κυβερνήσεις των χωρών των Βαλκανίων που είναι υποπροσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διαδοθεί ιδιαίτερως η έκθεση αυτή στις, σε αυτές τις χώρες καθεαυτές, την χάνει ευρεία ανάγνωση και ελπίζουμε ότι θα μας βοηθήσει η έκθεση αυτή τα θέματα των γυναικών να ξαναμπούν ψηλά στο κατάλογο προτεραιοτήτων ε, κατά τη ε, διαδικασία των, της προσχώρησης. Τροπολογία 6. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Άφετε 7. Ψηφοφορία κατά τμήματα. Είναι κανείς κατά αυτής της πρότασης. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική ένα Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δώδεκα Τροπολογία. Προφορική. αδιαφωνεί κανείς με την ε, πρόταση προφορικής τροπολογίας. Όχι, την ψηφίζουμε τότε υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 11. Ψηφοφορία κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 20 της άφετ υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Προχωρούμε. 9 της άφετ. Τμήμα 1. Υπέρ κατά Καταπίπτουν οι 13, 28, 23 και το δεύτερο τμήμα της 9 της ΑΦΕΤ. Όχι, ψηφίζουμε το ΑΦΕΤ 9, το τμήμα 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Οκτώ της ΑΦΕΤ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έντεκα της ΑΦΕΤ τμήματα ένα και δύο, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική τέσσερα, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε τώρα στην 5 της ΑΦΕΤ γιατί οι τρεις δεν ψηφίζεται η τρία δεν ψηφίζεται. Η πέντε λοιπόν της άφετη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δώδεκα της άφετ τμήμα 2-2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική πέντε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 19 τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Επομένως 25 και 15 της ΑΦΕΤ καταπίπτουν, 13 της ΑΦΕΤ υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Άρα πάμε στην 21 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 24 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 26 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. Να επαληθεύσουμε την 26. Άρχεται η ψηφοφορία και θα κλείσει λίγαν συντόμως. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. «27 υπέρ» κατά, αποχές, εγκρίνεται. 29 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 6 της άφετη υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 30 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 19 καταπίπτει. 31 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 32 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεν ψηφίζεται η μία τη ΑΦΕΤ, οι δύο τη ΑΦΕΤ. Ποιο είναι υπέρ. Κατά Αποχέ. εγκρίνεται. 33 υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. 34 υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. 36 υπέρ. Κατά απόχέ εγκρίνεται. 10 τη άφετ υπέρ. Κατά απόχέ εγκρίνεται. Συμβιβαστική 8 υπέρ. Κατά απόχέ, εγκρίνεται. Άρα ψηφίζουμε την 38 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 39 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 40 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 9 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε τώρα στην 41 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται.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 14-14 υπέρ και κατά. 51 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 52 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 8 υπέρ. Κατά. Συμβιβαστική 8 υπέρ. 10 του λένε του Προέδρου. Ναι, αλλά 8 γράφει το χαρτί. στο δικό μου έγγραφο είναι συμβιβαστική 8. Καλώς, είναι τυπογραφικό λάθος, θα έπρεπε να είναι συμβιβαστική υπαριθμών 10. Είναι η συμβαστική τροπολογία για την ενδέκατη παράγραφο του κειμένου, επομένως είναι η συμβαστική τροπολογία υπαριθμών 10, παρόλο που στο δικό μου χαρτί ε, γράφει 8. Αυτήν λοιπόν ψηφίζουμε. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Να ρωτήσω λοιπόν το εξής. Από την 55 μέχρι την 76 μπορούμε να τις ψηφίσουμε on block όλες μαζί. Αλήθεια μου λέτε. Υπάρχει κανείς που δεν θέλει. Εντάξει. Τότε 55 με 69. Μπορούμε 55 με 69 να τις ψηφίσουμε αν block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 67-68 απορρίπτεται. 68-69 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 70 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 71 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 72 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 19 υπέρ. Συγγνώμη λέει ο πρόεδρος. 73. 73 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 74 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 75 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 76 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται να το επαληθεύσουμε την 76 ψηφίζουμε ηλεκτρονικά ξεκινάει η ψηφοφορία τέλος της ψηφοφορίας εγκρίνεται και αυτή 77 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Να την επαληθεύσουμε. Ξεκινάει η ψηφοφορία για την 77. Τέλος της ψηφοφορίας. Δεν έχει σημασία, εγκρίνεται. 17 προς 11, μία ε, υπερβολική για τους σοσιαλιστές. Τέλος πάντων, πάμε στην 79. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 78 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 80 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 81 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 82 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 83 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 84 υπέρ. Κατά αποχές να το επαληθεύσουμε ηλεκτρονικός. Ξεκινά η ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 84. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται για μία ψήφο. 85 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 86 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 88 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 87 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Μπορούμε να ψηφίσουμε μαζί από το 89 ως 2, unblock, όχι. Καλά. 89 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 90 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 91 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 92 υπέρ. 92 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 93 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 94 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 95 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Από εδώ και πέρα μπορούμε να τις ψηφίσουμε μαζί. Ούτε τώρα. Εάν έστω και ένας λέει όχι, το δεχόμαστε. 96 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 97 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 98 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 99 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 100 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 101 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 102 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3 υπέρ κατά από εγκρίν, απορρίπτεται. Να το ελέγξουμε, ναι, ψηφίζουμε την τροπολογία υπαριθμό 3, ξεκινάει η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας, απορρίπτεται. Πράγματι απορρίφθηκε, 15 κατά 13 υπέρ. Να το ξαναδούμε. Ξαναψηφίζουμε την 3. Ξεκινάει η ψηφοφορία για την τροπολογία περιθμών 3. Τέλος. Απορρίπτεται 15 κατά, 13 υπέρ. 4 τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 5 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 1 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 2 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Πάμε τώρα το σύνολο του ψηφίσματος. Ξεκινάει η ψηφοφορία για το συνολικό κείμενο. Πέρας. Εγκρίνεται σαφέστατα συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Πάμε στο σημείο... Α. Πάμε στο σημείο 10. Αναπτυξιακή στόχη τη χιλιετία, ορισμό του πλαισίου μετά το 2015. Η συγγήτρια θέλει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω του συναδέλφου, του κοιόδη εισηγητέ που μου επέτρεψαν να εμπλουτίσω αυτή την έκθεση. Το κείμενο που θα ψηφίσουμε σήμερα είναι φιλόδοξο, που εστιάζει σε κάποιε πτυχέ. Ε, μία τεχνική παρατήρηση. Δεν ε, θέλω να υποστηρίξετε την 19 και 43 τροπολογίες όχι για λόγους ουσίας, αλλά για λόγους διάρθρωσης και συνέπειας με το συνολικό κείμενο. Δηλαδή, αν ψηφιστούν αυτές οι τροπολογίες, όλη η δομή της έκθεσης θα αλλάξει. Δεύτερη παρατήρηση για την τροπολογία 53 και την χωριστή ψηφοφορία που η ECR και η GUE επιθυμούν. Δεν θα υπάρξουν τρεις, τρία τμήματα να ψηφίσουμε, γιατί το δεύτερο που αφορά τη λέξη καταναγκαστικό δεν υπάρχει στο αρχικό κείμενο και δεν θα ψηφιστεί. Επομένως, αυτό το δεύτερο τμήμα. Ευχαριστώ για την ε, ψηφοφορία αυτή κατά τμήματα που ζήτησε η Γκουε σε μία από τις μεταφράσεις α, μεταφράστηκε ως αναγκαστική πορνεία. Αλλά αυτό ε, δεν ε, υπήρχε στο αρχικό κείμενο. Θα έχουμε δύο τμήματα δηλαδή σε αυτή την ψηφοφορία. Έτσι. Το καταλάβαμε όλοι. Κυρία Παρβάνοβα, θέλει το λόγο. Ευχαριστώ. Μετά από αυτά που είπε η συγγήτρια για την τροπολογία 43, θέλω να διευκρινίσω κάποια πράγματα για την τροπολογία μου. θα πρέπει να αναφερθεί εκεί όχι η παράγραφος 4, αλλά η παράγραφος 4H. Δεν θέλουμε, θέλουμε να, να γίνει αυτή η μικρή αλλαγή, δεν θέλουμε να αλλάξει η αρχική παράγραφος 4. Ελπίζω να το κατάλαβαν όλοι. Και θα ζητήσω να δούμε μήπως κάποιος απορρίπτει την προφορική τροπολογία ε, και αν το απορρίπτει δεν θα μπορέσουμε να την ψηφίσουμε, αλλά θα το ρωτήσουμε να φτάσουμε εκεί. Συμβαστική 1. Υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείτε. Τροπολογία 14. Υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείτε. Τι λέτε. νομοθετείτε δεν χρειάζεται να λέτε ε, κατά και τα λοιπά. Ε, όχι, είναι τμήμα της διαδικασίας. Πρέπει να δώσω στον κόσμο τη δυνατότητα να πει όχι εφόσον μπορεί και να θέλει. Αν βλέπω ότι όλοι ψηφίζετε υπέρ, δεν θα χρειάζεται να πω ε, κατά και αποχές. Αλλά αν όχι πρέπει να το πω για να δώσουν ευκαιρία να καταψηφίσουν. 15. Υπέρ, κατά, αποχές. Δεν είναι ασαφές. Ξανά. Υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται. 16. Υπέρ, κατά, αποχές. Υιοθετείται. 17. Υπέρ, κατά, αποχές. Ας το ελέγξουμε. Ας ελέγξουμε τη 17. Αρχίζει η ψηφοφορία ηλεκτρονικά παρακαλώ. Είχε υπερψηφιστεί με δύο ψήφου επιπλέον. Συμβασμό 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείται. Τροπολογία 19. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 20. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 21. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείται. Η 22 καταπίπτει. Πάμε στην 23 με, με ψηφοφορία κατά τμήματα. Το πρώτο τμήμα της προφορής κατά τμήματα της τροπολογίας 23. Υπέρ, κατά, αποχές. Θα το ελέγξουμε γιατί δεν ήταν σαφές. Πρώτο τμήμα της 23. Ψηφίζουμε τώρα. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται με δύο ψήφους κατά, παραπάνω. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογή 24 υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται. 25 αποσύρεται, 26 υπέρ, κατά αποχές, υιοθετείται. Ελέγχουμε την 26. Ψηφίζουμε τώρα την 26. Πέρας ψηφοφορίας. Υιοθετείται. 53. Είναι ψηφοφορία κατά τμήματα. Δεν θα είναι τρία τμήματα όπως είπαμε, αλλά δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείτε. Η 42 καταπίπτει. Η 32 καταπίπτει πιο σωστά. Πάμε στην 27. Είναι προφορική α, τροπολογία. Υπάρχει αντίρρηση, όχι. Την ψηφίζουμε λοιπόν. Υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείτε. 28. Υπέρ, κατά, αποχές Υιοθετείτε. 29 υπέρ κατά αποχές Υιοθετείτε. 30 υπέρ κατά αποχές Υιοθετείτε. 31 υπέρ κατά αποχές Υιοθετείτε. 33 υπέρ κατά αποχές Υιοθετείτε. 34 υπέρ κατά αποχές Υιοθετείτε. Συμβασμός 3 υπέρ κατά αποχές 36 υπέρ κατά αποχές υιοθετείτε, 38 υπέρ κατά αποχές υιοθετείτε, 39 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται, 40 υπέρ κατά αποχές υιοθετείτε, 41 υπέρ κατά αποχές υιοθετείτε, 42 υπέρ κατά αποχές υιοθετείτε και πάμε στις 43 που είναι προφορική τροπολογία. Υπάρχουν αντιρρήσεις να την ψηφίσουμε αυτή την προφορική τροπολογία. Όχι. Την ψηφίζουμε λοιπόν. Υπέρ. Κατά. αποχές Υιοθετείτε. Οι 44-45 λοιπόν καταπίπτουν και ψηφίζουμε τη 46. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. 47 υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. 49 υπέρ. Κατά αποχές υιοθετείται 50 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται 51 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται 52 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται 54 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται 55 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται 56 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται 57 κατά αποχές υιοθετείται απορρίπτεται, 58 υπέρ, κατά αποχές υιοθετείται, 59 υπέρ, κατά αποχές δεν κατάλαβα, το ελέγχουμε. Ελέγχουμε την 59. Ψηφίστε τώρα ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας. Σαφώς υιοθετήθηκε. 60 υπέρ κατά αποχές υιοθετείτε. 61 υπέρ κατά αποχές υιοθετείτε. 6 είναι προφορική τροπολογία. Υπάρχει αντίρρηση να την ψηφίσουμε. Όχι. Ψηφίζουμε την 6 υπέρ κατά αποχές υιοθετείτε. 7 υπέρ κατά αποχές υιοθετείτε. 8 υπέρ 9 α, απο, αποχε, κατά Υιοθετείτε 9 υπέρ κατά αποχές υιοθετείτε. 1 υπέρ κατά αποχές υιοθετείτε. 2 υπέρ κατά αποχές υιοθετείτε. 3 υπέρ κατά αποχές υιοθετείτε. 4 υπέρ κατά αποχές υιοθετείτε. Άρα η 5 καταπίπτει. Ψηφίζουμε όλο το ψήφισμα. Ψηφίστε τώρα. Πέρας προφορίας. Υιοθετείτε. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Και τώρα πάμε στο επόμενο σημείο πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ταμείο Ενίσχυσης των Απόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ζητήσω από την εισηγήτρια αν θέλει να πάρει το λόγο. Όχι, δεν θέλω. Όχι, δεν θέλετε. Και τώρα θα ξεκινήσουμε τις ψηφοφορίες. Τροπολογία 56. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. 57. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβασμός 4. Υπέρ κατά, αποχές υιοθετείτε 12 υπέρ, κατά, αποχές υιοθετείτε. Συμβασμός 5 υπέρ, κατά, αποχές υιοθετείτε. 64 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 65 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 14 υπέρ, κατά, αποχές υιοθετείτε. 66 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 67 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. Συμβασμός 6 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. 68 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. Συμβασμός 7 υπέρ. Θέλετε να ελέγξουμε την 68. Παρακαλώ. Ηλεκτρονικά ψηφίστε τώρα. Πέρας ψηφοφορίας. Υιοθετείτε. Συμβασμός 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Τροπολογία 71. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Θέλετε να ελέγξουμε την 71. Ψηφίστε τώρα ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας είχε απορριφθεί με μία ψήφο διαφορά. Δεν το είχα δει. Συμβασμός 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. 18. Υπέρ. Κατά. Αποχές. υιοθετείτε. 75. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 74. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά την 74. Ψηφίστε τώρα. Απορρίπτεται. 19. Καταπίπτει όμως. Πάμε στην 76. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβασμός 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Διοθετείται. 21. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 80. Θέλετε να ελέγξουμε την 21. Ψηφίζετε τώρα ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 80. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 22. Και 77 που είναι ίδιες. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετούνται. Η 23 καταπίπτει. Πάμε στην 81. 81 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 24 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 82 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 83 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 25 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έχουμε την 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 86 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 87 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 28 καταπίπτει, 30 αποσύρεται, 89-90 ταυτόσημες, υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετούνται. Ελέγχουμε τις 2, 89 και 90 ηλεκτρονικά, ταυτόσημες. Άρχεται η ψηφοφορία, πέρας της ψηφοφορίας. Α, απορρίπτονται. 91, υπέρ, κατά, αποχές, Απορρίπτεται 92, 93, 94 ταυτόσιμες. Υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτονται 95 υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται 31 υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. 97 υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. 96-98 κατά πίπτου. 99 υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνονται. Εγκρίνεται 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 107-108 ταυτόσημες υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. Ηλεκτρονικός έλεγχος 107-108. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Απορρίπτονται. Τριάντα τέσσερα, υπέρ, κατά, αποχές, Νομίζω εγκρίνεται. Αλλά ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά τη 34. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 33. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 109. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος. 109. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 1. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 37. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 2. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 38 κατά πίπτη. Τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 40 είναι ε, ψηφοφορίες ε, τμήματα. Το πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές Συγγνώμη, λέει ο πρόεδρος. Παναλαμβάνω. Πρώτο τμήμα. Υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται. 41. Υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. 42. Προφορική τροπολογία. Υπάρχει αντίρρηση στην ε, υιοθέτηση. Όχι. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 44 κατά πίπτη, 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το 5 καταπίπτει. 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 50 είναι ε, διαχωριστική σε δύο τμήματα. Το πρώτο εγκρίνεται, το δεύτερο υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Θα ελέγξουμε το δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 50 ηλεκτρονικά παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 7 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. 51 υπέρ κατά αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος. 51. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται ε, συμβαστική τρία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ξεχωριστή ψηφοφορία στο 9. Πρώτο τμήμα εγκρίνεται, δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 55 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ψηφίζουμε ολόκληρο το κείμενο όπως τροποποιήθηκε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα τη ψηφοφορία. Και υιοθετήθηκε συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Ε, we then had the last vote, and that's about the, uh, on social housing in Europe. Yeah, το, η επόμενη ψηφοφορία είναι η κοινωνική στέγαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελε η εισηγήτρια να μιλήσει. Πολύ σύντομα θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους και όλους τους εισηγητές, εισηγήτριες για την εξαιρετική εργασία την οποία κάναμε επί τη βάση όλων των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που ανταλλάξαμε. Έχουμε την τελική ψηφοφορία και ελπίζουμε να δικαιωθούμε. Έχουμε ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Okay, we start with compromise 4. Αρχίζουμε με τη συμβιβαστική 4 υπέρ κατά αποχές ε, υιοθετήθηκε 26 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται 29 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται 30 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται Συμβαστική 5 υπέρ, κατά, αποχές ε, υιοθετείται. Συμβαστική 6 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ, κατά, αποχές υιοθετείται. Συ... Ε, τροπολογία 41 είναι προφορική, υπάρχει αντίρρηση, όχι. Ωραία, ψηφίζουμε τη 41. Υπέρ, κατά, αποχές υιοθετείται. Και πάμε στην 38, σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, ε, απορρίπτεται. Συμβαστική 42, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 39, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 55 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 57 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 59 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 4 5 ε, συγγνώμη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τροπολογία 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 24 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ την 24. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 25 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το τροποποιημένο κείμενο, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας Εγκρίνεται σαφώς, υιοθετήθηκε λοιπόν συγχαρητήρια στην συγγήτρια. So we don't take 15 minutes break. Κάνουμε ένα διάλειμμα 15 λεπτών πριν ξεκινήσουν οι συντονιστές. Ευχαριστώ πολύ.